Colleagues, I think we can start. μπορούμε να αρχίσουμε νομίζω. Έγκριση της ημερήσιας. Παρακαλώ. Ένα διαδικαστικό έχω. Θα ήθελα να μου δοθεί μια εξήγηση γιατί αναβλήθηκε το σημείο σε σχέση με την ετήσια έκθεση απάντηση αναβλήθηκε διότι όπως ξέρετε η ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο Μοσκοβίση ήταν να γίνει ε, την περασμένη εβδομάδα αλλά το αναβάλαμε διότι ο κ. Γιούνκερ ανέβαλε την εξαγγελία την ε, παρουσίαση μόνο που αναμενόταν να κάνει ο κύριος Μουσκοβησής στην Επιτροπή μας. Είχαμε προσπαθήσει αρχικά να εγγράψουμε το σημείο στη σημερινή συνεδρίαση. Πολλά μέλη της Επιτροπής όμως ε, θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να γίνει το βράδυ σε μια έκτακτη συνεδρίαση δηλαδή της Επιτροπής ΕΚΟΝ, αλλά έπρεπε να εγγραφεί σε μια τακτική συνεδρίαση. Η μοναδική δυνατότητα λοιπόν ήταν η αυριανή ημερομηνία. Συμφωνήσαμε όμως με τον εισηγητή να αναβληθεί η συζήτηση για τις 15 επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό και είχαμε αυτή την αναβολή κατά μία εβδομάδα. Δεν θα επηρεαστεί όμως ο σχεδιασμός στο χρονοδιάγραμμα της έκθεσης. Ε, η κυρία Σκοτράτο, ε, με ανησυχεί αυτό διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα λάξε λήξε. Καταλαβαίνετε ότι μας απασχολεί όλους πάρα πολύ το ταχύτερο δυνατόν επιθυμώ να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή. Όπως σας έλεγα, ε, στις 15 έχουμε τη συζήτηση για την έκθεση για τη φορολογία. Στη συνέχεια, η διάσκεψη των Προέδρων αναμένεται να λάβει απόφαση σχετικά με την ε, απάντηση που θα δώσει το Κοινοβούλιο γενικότερα για τα φορολογικά ζητήματα. Κάποιοι ζητούν εξεταστική επιτροπή, άλλοι διαφωνούν. Η διάσκεψη των Προέδρων αυτή την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, θα αποφασίσει και με γραπτή διαδικασία ακόμη νωρίτερα. Όμως αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε την ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου για τα φορολογικά ζητήματα και η διάσκεψη των Προέδρων θα πάρει την απόφαση για την στάση που θα τηρήσει το Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι έχει οθετήσει προς ανατολισμό η Επιτροπή ΕΚΟΝ, αλλά την τελική απόφαση θα την πάρει η Διέσκεψη των Πρόεδρων. Κ. Λάγκεν. Παρατήρηση θέλω να κάνω. Μια παρατήρηση για τις συναντήσεις με τον κύριο Μοσκοβισή. Δευτέρα βράδυ 9 9.30 ε, είναι το ίδιο άβολο όπως και απόψε. Έχουμε αρκετό χρόνο για κανονικές συνεδριάσεις που τέλειωναν κανονικά νωρίτερα. Και σας παρακαλώ λοιπόν, Πρόεδρε, και σας συνεργάτες, τέτοιου είδους χρονικές ε, στιγμές, σε τέτοια, ε, με τέτοια καθυστέρηση ώρα, να μην επαναληφθούν. Να βολεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογα με το δικό μας ωράριο. Ευχαριστώ. Uh, uh, ναι, ε, σημειώσαμε την ε, θέση κάποιων ομάδων και γι' αυτό το προβλέψαμε για αύριο το πρωί, όχι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί. Λοιπόν, θεωρώ ότι εγκρίνουμε έτσι το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Πρώτον, ε, κοινή συνεδρίαση την Τρίτη στις 8 ανάμεσα στην Επιτροπή ΣΕΚΟΝ και ε, Απασχόλησης. Παρουσία των ε, Ντομπρόφσκι, Μοσκοβισή και Τάισεν για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης και το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και θα συζητηθεί το θέμα του οικονομικού, θεσμικού οικονομικού διαλόγου και των επιπτώσεών τους. μόλις ολοκληρωθεί η σημερινή συνεδρίαση θα ορίσουμε την αίθουσα που θα διεξαχθεί η κοινή συνεδρίαση αυτών των επιτροπών. Δεύτερον, ενέως εποπτικός μηχανισμός, οι, συντονισμοί, οι συντονιστές συγγνώμη, στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισαν να γίνουν τρεις ακροάσεις το 2015 με τον πρόεδρο του Συμβουλίου ε, εποπτείας και δύο, βασι... δύο ακροάσεις ε, που προβλέπονται από ε, την Διαθεσμική Συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στις 31 ε, Μαρτίου του 2015 θα γίνει η πρώτη έκτακτη ακρόαση. Ε, η πρώτη τακτική ακρόαση ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και η δεύτερη θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου του 2015. Για τους τριμερείς ε, διαλόγους έχουμε πολύ καλά νέα. Στις 26 ε, Νοεμβρίου η διαπραγματευτική ομάδα σε συνεργασία με την Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό που θεσπίζει τα σε τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία Επετεύθη η συμφωνία παρουσία του Επιτροπού Τζόναθαν Χιλ. Θα ήθελα να συγχαρώ τη διαπραγματευτική ομάδα του, ε, της ΕΚΟΝ και κυρίως τον κύριο Λαμασούρ. Ξέρετε ότι πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, μες όχημα, για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και έτσι θα συμβάλλει το Κοινοβούλιο στο επενδυτικό πρόγραμμα των 315 δισεκατομμυρίων του, του κυρίου Γιούνκερ, δηλαδή αναδεικνύονται σε προτεραιότητα αυτά τα έλλειψη στο επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. θα διατηρηθεί το χαμηλότερο όριο των 10.000 ευρώ για τις λιανικές αν θέλετε επενδύσεις αλλά τα έλτιψε θα προστατεύουν την αποπληρωμή της ε, περαιτέρω υποχρεώσεις για τη θέση σε εμπορία για τους ε, κατόχους των νέων χρηματοδοτικών μέσων, όρους λειτουργίας των έλτιψε και φυσικά θα γίνει διαβούλευση με την ΕΚΟΝ όπως προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση του κειμένου. Για την οδηγία κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος έγινε επίσης στο Στρασβούργο η τελευταία συνεδρίαση είναι κοινή ορμοδιότητα βάσει του άρθρου 55 με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και συζητούμε ακόμη βασικά ζητήματα όπως η προστασία των δεδομένων, αποτίμηση κινδύνου και πολλά άλλα συναφή ζητήματα. Επόμενος τριμερής θα γίνει την 3η στις 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα και είμαστε σε επαφή με τη διαπραγματευτική ομάδα της Επιτροπής ΕΚΟΝ για να επιτύχουμε κάποια βήματα προόδου στα πλαίσια του τριμερούς αυτού διαλόγου. Ολοκληρώνω έτσι τις ανακοινώσεις και μπορώ να περάσω στην ακρόαση για τον διορισμό του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής, ΕΣΚΑΠ. Δημόσια ακρόαση με τον κύριο Μάρτι Χετεμάκη. Σας καλωσορίζω είστε ο Υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομικών της Φιλανδίας και ε, από το 2003 ως το 2013 ήσασταν αντιπρόεδρος του EFC και ασχολούσασταν ακριβώς με τα στατιστικά ζητήματα. Ε, ξέρετε ότι βάσει το κανονισμό 235 του 2008 το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει έναν υποψήφιο και το Κοινοβούλιο θα ε, κληθεί να εγκρίνει τον υποψήφιο για τον ΕΣΚΑΠ, για αυτό τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα λοιπόν την πρόταση για τον κύριο Μάρτι Χετεμάκη και θα αρχίσει η επίσημη δημόσια ακρόαση ε, του κυρίου Χετεμάκη. Ε, θα έχετε ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή σας για την αρχική παρουσίαση και μετά θα αρχίσουν οι ερωταπαντήσεις όσοι Παρακαλούμε, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή για την πρόσκληση να είμαι ενώπιόν σας. Στις πολύ σύντομες παρατηρήσεις μου θα επικεντρωθώ πώς βλέπω τον ρόλο της ΕΣΓΑΜ. Πρώτα, θέλω να υπενθυμίσω τους λόγους που οδήγησαν στην συγκρότηση, στην δημιουργία της ΕΣΓΑΜ. Το Νοέμβριο 2005 το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ συνεπέρανε ότι ένα υψηλού επίπεδου όργανο θα αύξανε την ανεξαρτησία και την λογοδοσία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Τότε ήμουν μέλος της Οικονομικής ε, ε, Επιτροπής ε, και προέδρευα της Επιτροπής Στατιστικών. Υπό αυτή μου την ιδιότητα εργάστηκα για να συγκροτηθεί η ΕΣΓΑΜ. Ο άμεσος λόγος για τη συγκρότηση της ΕΣΓΑΜ ήταν τα λανθασμένα στοιχεία, στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας και τότε υπήρχαν και γενικότερου χαρακτήρα επιχειρήματα για αυτό τους λόγους. Για τρεις λόγους σημαντικούς ήταν σημαντικό να υπάρχει κοινό κώδικας πρακτικών όσον αφορά τις στατιστικές αρχές και ένα σώμα που θα αξιολογούσε και θα ανέφερε σε σχέση με τα της εφαρμογής αυτού του κώδικα. Αυτοί οι τρεις λόγοι εξακολουθούν να έχουν ισχύ σήμερα, να είναι ισχυροί. Ο πρώτος λόγος ε, για τον κώδικα και την ΕΣΓΑΜ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα. Πόσο δηλαδή, σε ποιο βαθμό οι πολιτικές βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία. Για τα έσοδα, για παράδειγμα, συλλέγονται με βάση τα εθνικά στατιστικά στοιχεία, καθώς επίσης και για τις δαπάνες. Πολλές φορές βασίζονται σε στατιστικά στατιστικά στοιχεία των εθνικών αρχών και επιπλέον οι οικονομικοί κανονισμοί εποπτεύονται για την υλοποίησή τους με βάση πάντα στατιστικά στοιχεία. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια χώρα όπου τα στατιστικά στοιχεία να διαδραμάτιζαν ένα τόσο σημαντικό ρόλο στην λήψη πολιτικών αποφάσεων. Μια και έχουν τέτοια σπουδαιότητα τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε σαφής ανάγκη να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα αυτών των στοιχείων απαιτώντας από τις στατιστικές αρχές να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές υψηλού επίπεδου σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο δεύτερος λόγος για τον κώδικα πρακτικών και την ΕΣΚΑΠ είναι τα, η εμπιστοσύνη στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι αυτή η εμπιστοσύνη τόσο υψηλού επίπεδου όπως θα έπρεπε. Πέρυσι το Κοινοβούλιο εξέτασε σε σχέση με, μια κράτη, με μια, ένα κράτος και συνέταξε μια αναφορά για τα, την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων αυτής της χώρας. Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου αναφερόταν σε μια μελέτη επιπτώσεων και σύμφωνα με είναι, η εμπιστοσύνη ήταν πολύ χαμηλή. Ερωτήθηκαν οι ε, πολίτες αν ε, τα στατιστικά στοιχεία παράγονται χωρίς επίσημη ανάμειξη και συμφωνεί μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή η πλειοψηφία δεν θεωρεί ότι ε, σε σχέση με αυτά τα στοιχεία είναι ελεύθερα πολιτικής ε, επιρροής. Παρότι αυτά τα αποτελέσματα αναφερόντουσαν σε μια χώρα θέλω να πω ότι ανεπαρκής εμπιστοσύνη στα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι ένα πιο γενικό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή έχει κέριο χαρακτήρα ε, ο ρόλος των στατιστικών στοιχείων για την πολιτική και την λήψη αποφάσεων. Δεν μπορεί να αναμένει κανείς ε, πολίτες να έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές πολιτικές όταν ε, δεν έχουν εμπιστοσύνη σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία με βάση τα οποία αποφασίζονται και λαμβάνουν αποφάσεις για αυτές πολιτικές. Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι ανεπάρκειες των στατιστικών στοιχείων δεν αφορούν μόνο κάποιες λίγες χώρες. Ουσιαστικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει πολλά να πράξουν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κώδικα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, οι ε, απαιτούμενες βελτιώσεις ε, δεν απαιτούν πρόσθετα κονδύλια ή μεγάλες διοικητικές προσπάθειες. Πράγματι μεγάλη πρόοδος έχει ήδη επιτευχθεί και παραμένουν αρκετά να γίνουν. Όταν ο κώδικας πρακτικών προετοιμάστηκε έγινε κάποια συζήτηση αν θα έπρεπε να έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν θα ήταν ευκταίο να ρυθμιστούν οι πρακτικές αρχές των εθνικών στατιστικών αρχών. Η ήπια προσέγγιση με την ήπια νομοθεσία που υιοθετήθηκε υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εξέτασης των ομοτήμων στατιστικά υπευθύνων και ο ρόλος που έχει η ΕΣΚΑΠΑ για να αναφέρει τα σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι δεδομένος. Είχα μια ευκαιρία με την ΕΣΚΑ πριν από έξι χρόνια να ασχοληθώ με αυτά. Η πρώτη ομάδα δημιουργήθηκε στη νέα δομή της, ε, του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και η πρώτη έκθεση του 2009 ταυτοποίησε, εντόπισε κάποιες αδυναμίες, πρώτες αδυναμίες σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία για παράδειγμα σε σχέση με την πρόσληψη και την απόλυση επικεφαλής υπηρεσιών στατιστικών ε, στα κράτη-μέλη. Και επέμεινε ότι για αυτές τις διαδικασίες ε, θα πρέπει να παραμένουν αυτές ανεξάρτητες από την πολιτική εντολή και πολιτική ανάμειξη. Η ομάδα σε σχέση με την ΕΣΓΑΠ πρόσφατα έκανε μια εξέταση και ανάλυση σε σχέση με την Eurostat. Σας υπευλήθη έκθεση πριν από λίγες εβδομάδες ε, από τον επικεφαλής. Είμαι υπέρ της στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΣΓΑΜΠΑ και Eurostat, σίγουρα. Η συνεργασία <clears throat> διευκολύνει το έργο της ΕΣΓΑΠ, ενώ ταυτόχρονα δεν περιορίζει την ανεξαρτησία της ΕΣΓΑΠ. Συμφωνώ λοιπόν με τις συστάσεις της ΕΣΓΑΠ όσον αφορά την Ευρωστάτ, όπως σας παρουσιάστηκαν από την τρέχουσα έκθεση. Ιδιαίτερα συνέστησε η ΕΣΚΑΠ ότι ρυθμίσεις για την πρόσληψη γενικού διευθυντή της Ευρωστάτ θα πρέπει να καθορίζονται νομικά και να βασίζονται σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό έτυχε να είμαι μέλος της ε, Επιτροπής Επιλογής σε σχέση με την διαδικασία επιλογής που ήταν πράγματι πολύ διαφανής και βασιζόταν σε μια πολύ προσεκτική αξιολόγηση των επαγγελματικών ικανοτήτων όσον αφορά τους υποψήφιους. Βασίζομαι στο ότι μια παρόμοια διαδικασία θα υιοθετηθεί και θα ισχύει στο μέλλον. Όμως θεωρώ ότι είναι ενδεδειγμένο να βελτιώσουμε την εφαρμογή των αρχών όσον αφορά την πρόσληψη αυτών των υψηλά ισταμένων υπαλλήλων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δύο λόγια στο τέλος σε σχέση με α, τις δράσεις της Επιτροπής. Συμφωνώ με την Προεδρία της ΕΣΓΑΠ ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι σημαντικός και ισχυρός εταίρος και σύμμαχος της ΕΣΓΑΠ. Θα ήθελα να υποβάλω μια ιδέα να εξεταστεί από την ε, δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚΟΝ ότι ο κώδικας πρακτικών είναι ένα μέσο ήπιας νομοθεσία νομοθεσίας που η αποτελεσματικότητα της, αυτής της διαδικασίας βασίζεται στον δημόσιο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, όσον αφορά κάτι το σημαντικό σε ένα κράτος μέλος ε, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να μην είναι ανάγκη μια διορθωτική ε, κίνηση. Ωστόσο όμως θα έπρεπε από την Επιτροπή να υπάρξει η αναγκαία δράση για την ενημέρωση και την αναγκαία λογοδοσία. Πράγματι, ακόμα και η δυνατότητα μιας τέτοιας ακρόασης από την Επιτροπή ΕΚΟΝ θα μπορούσε να είναι αποτρεπτικό, ισχυρό αποτρεπτικό συστοιχείο ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές πρακτικές. Γενικά, η δημόσια προσοχή που μπορεί να επιτευχθεί μπορεί να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα ώστε να αποφεύγονται όλοι στήματα στο μέλλον. Για να υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τα μέλη της Επιτροπής θα ολοκληρώσω εδώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χετεμάκη για τη δήλωσή σας, καθώς επίσης και για την πρότασή σας, την οποία θα λάβουμε δεόντως υπόψη. Και αν κατάλαβα καλά, Ε, μπορεί να πρέπει να χρειάζονται κάποια τυπικά ζητήματα για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή μας το δικαίωμά της ε, για να ε, το συσχετίσουμε και με τις διαδικασίες ήπιας νομοθεσίας και δεν χρειάζονται νομικές διατάξεις. Είναι μια καλή ιδέα αυτή, την οποία θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Μπάλτς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Δύο ερωτήσεις έχω να σας θέσω. Στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βιώσαμε πόσο σημαντικά είναι τα στατιστικά στοιχεία, ε, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως και να είναι και ακριβή και κυρίως να είναι συγκρίσιμα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγα περισσότερα για τη συνοχή των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων και πού ε, έγινε η βασική ευθύνη κατά την άποψή σας για αυτά τα συνεκτικά στατιστικά στοιχεία. Δεύτερη ερώτηση. Στην ετήσια έκθεση λέγεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ε, η ανεξαρτησία ε, στατιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ε, δεν είναι γενείς ε, σε, αυτά τα, ε, σε αυτές τις στατιστικές υπηρεσίες. Θεωρείτε εσείς ότι δεν υπάρχει επαρκής ανεξαρτησία σε αυτές τις στατιστικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Χιτερμάκη. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ κύριε Μπάλς για την ερώτηση. Για να απαντήσω στη δεύτερη ερώτησή σας για το κατά πόσον υπάρχουν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχουν ε, απτές αποδείξεις θα έλεγα για την επιρροή πολιτικών αρχών στα επίσημα στατιστικά στοιχεία, αλλά συχνά υπάρχουν κάποιες ε, συμπτώσεις, για παράδειγμα, στην αλλαγή κυβέρνησης και στην αλλαγή του επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Και αυτό Φυσικά μπορεί να δημιουργήσει υποψίες ότι κάποια σχέση υπάρχει και υπάρχει πολιτική παρέμβαση. για τα στατιστικά στοιχεία. Και αυτό επανέρχεται στην πρότασή μου. ο φόβος της δημόσιας ακρόασης μπορεί να αποτελήσει σημαντικό ανασταλτικό παράδειγμα ε, για παρέμβαση στα στατιστικά στοιχεία. Ε, σε μια χώρα υπάρχει μια υπόθεση που εκκρεμεί όσον αφορά το ρόλο του επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας, ο οποίος ε, αυτή τη στιγμή διώκεται ποινικά. Υπάρχει όμως μια νομική διαδικασία και πολύ δύσκολα φυσικά μπορεί να την επηρεάσει κάποιος έξωθεν. Εδώ αναφέρομαι στον επικεφαλής της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας. Στην πρώτη σας ερώτηση τώρα, όσον αφορά τη συνοχή των στατιστικών στοιχείων, η ουσία είναι να είναι συγκρίσιμα τα στατιστικά στοιχεία ε, των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει κάπως να καλυφθούν. Παραδείγματος χάρη στον τομέα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων, κάθε χρόνο υπάρχει μια ετήσια έκθεση για την πρόοδο των διαφόρων στοιχείων στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ. ε, σύντομες ερωτήσεις παρακαλώ από τους αδέλφους γιατί αλλιώς δεν θα μας φτάσει ο χώρος για ερωτήσεις και απαντήσεις. Από πλευρά Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο κύριος Μπαγιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Χετεμάκη που έχετε έρθει εδώ σήμερα και καλή επιτυχία για την πιθανή μελλοντική σας αποστολή ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Ε, είστε εταίρος φυσικά της Επιτροπής ΕΚΟΝ και κατά την άποψή σας ποια είναι τα ισχυρά και τα ε, σημεία και οι αδυναμίες και πώς θέλετε να διαχειριστείτε το Συμβούλιο αυτών των στατιστικών υπηρεσιών. Ο συνάδελφό μου αναφέρθηκε στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων και ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο ασχολείται με το θέμα του κανονισμού 223 και τίθεται λοιπόν και το εξής ερώτημα. Ε, τι γίνεται με την πολιτική ε, παρέμβαση για τους ε, διευθυντές και της Eurostat, των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, αλλά και της Eurostat. Πώς μπορούμε να έχουμε ανεξαρτησία σε σχέση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και την άποψή σας από αυτού. Θεωρείτε ότι η ανεξαρτησία της Eurostat είναι κάτι δεδομένο, πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το διευθυντή. Ο διευθυντής της Eurostat είναι ουσιαστικά και ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών λοιπόν θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε είναι άμεσα υπόλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κώδικας ε, καλών πρακτικών που ίσως θα έπρεπε να δημοσιευθεί είναι πολύ καλή ιδέα κατά την απόψή μα, και, αλλά ακούμε και κάποια κράτη-μέλη όμως να μας λένε ότι εμείς θα θέλαμε περισσότερες ανταλλαγές απόψεων με το Κοινοβούλιο και τη Eurostat, διότι γνωρίζετε μέχρι ποιου σημείου είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε σε κάποιους κανόνες και κάποιου ορισμού και εφαρμογέ στα στατιστικά στοιχεία. Και κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι η Eurostat πάντα δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν εισακούονται επακριβώ οι στατιστικέ υπηρεσίε των κρατών μελών και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται κυρίω με τι ακροάσει των στατιστικών υπηρεσιών και το ε, γεγονό ότι κατά πόσον η Eurostat είναι εταίρο και μπορεί να απαντά στι ερωτήσει των στατιστικών υπηρεσιών ε, όπω ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπεγέ. Πρώτα απ' όλα με ρωτήσατε για τα τροτά σημεία και για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ΕΣΚΑΠ, αν κατάλαβα καλά. Εγώ πιστεύω πως ε, επιρροή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν μιλάμε για τους ηθήνοντες ε, της ε, στατιστικής διακυβέρνησης τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη-μέλη. Δέχεται οι γνωμοδοτήσεις και οι εκθέσεις της ΕΣΚΑΠ να μην έχουν μεγάλο ειδικό βάρος αν δεν εισακουστούν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Πολλά εξαρτώνται από το αν θα εισακουστεί το μήνυμα που περνάμε. Παρότι το περιεχόμενο μπορεί να είναι καλό, το βασικότερο ζήτημα είναι πώς θα επηρεάσει τη τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής. Και αυτό, ξαναλέω, εξαρτάται από την υποδοχή που θα επιφυλάξει το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο ε, στις εκθέσεις μας και στις γνωμοδοτήσεις μας. Ε, τώρα, περνάω στη γύρω και το θέμα του κανονισμού. Νομίζω ότι το βασικό εδώ, ε, και αυτό τονίζεται και στον κώδικα, είναι η διαδικασία διορισμού και απομάκρυνσης ε, του επικεφαλής ε, της Eurostat. Η διαδικασία διορισμού φυσικά ε, πρέπει να είναι διαφανής, ανοιχτή και να βασίζεται στην επαγγελματική επάρκεια. Η Επιτροπή είμαι πεπισμένο θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτού του είδους τη διαδικασία επιλογής και διορισμού. συστήνων ανεπιφύλακτα να ε, καταγραφούν ε, στον κανονισμό ή σε κάποιο άλλο νομοθέτημα ε, οι αρχές που θα διέπουν αυτή τη διαδικασία. Θα είμαι πολύ σύντομος να απαντήσω και στο τελευταίο ερώτημα. σχέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Νομίζω τώρα έχουμε εγκαθιδρύσει ένα τρόπο επικοινωνίας, το peer review, αποτίμηση ομοτήμων, αρκετά επαχθής διαδικασία όπου η Eurostat αποτιμά ε, τις ε, πρακτικές ε, ως προς την εκπόνηση στατιστικών στοιχείων στα κράτη-μέλη. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρακαλώ να μην υπερβαίνετε το ένα λεπτό με τις ερωτήσεις σας, ε, διότι αν ε, υποβάλλετε ερωτήματα δύο λεπτών, ξυπακούεται ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος και για, την απάντηση και δεν έχουμε τόσο χρόνο. Κύριο Στανίσλαφ Ότσοκ από, τη, από τους συντηρητικούς. Panie Przewodniczący, Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πω ότι το εκτίμησα ιδιαίτερα την αξιόλογη αυτή και σύντομη παρουσία σας που επικεντρώνεται στα θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Και για τις ερωτήσεις έχω κάποιες ερωτήσεις. Σύμφωνα με εσάς, ο κώδικας πρακτικών είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα όσον αφορά τα στατιστικά ή θα έπρεπε να, βελτιωθεί περαιτέρω αυτός ο κώδικας μήπως θα έπρεπε να υπάρξει κάποια ε, επανεκπώνηση από την ΕΣΚΑΠ παίρνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι λειτουργούν αυτή τη στιγμή χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες πώς θα μπορούσαμε ουσιαστικά να πετυχαίναμε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά τα επίκαιρα στατιστικά στοιχεία πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων περαιτέρω δηλαδή Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο εσείς αποφασίσατε να υποβάλλετε αίτηση για αυτό το αξίωμα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θα πρέπει να βελτιωθεί ο κώδικας, θα έλεγα το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα του κώδικα αλλά πώς συμμορφώνονται οι διάφοροι υπεύθυνοι με αυτόν τον κώδικα. Και αυτό σχετίζεται με τη δεύτερη ερώτησή σας. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Και θα έλεγα επ' αυτού, όπως ε, είπα προηγούμενα, όλα, όλα τα κράτη-μέλη έχουν πολλά να πράξουν για να συμμορφωθούν με τα όσα επιτάσσει ο κώδικας αυτός. Και επίσης Ίσως θα μπορεί να υπάρχουν κάποια απλά πράγματα όπως οι διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης των επικεφαλής των στατιστικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων από τα κράτη-μέλη. Απλά πράγματα δηλαδή. Νομίζω όμως ουσιαστικά ότι μπορώ να πω ότι η επαγγελματική ακαιρεότητα και αξιοπιστία και ικανότητα όταν βελτιωθούν και μπορούν να βελτιωθούν, ε τότε θα, βελτιωθούν, θα βελτιώσουν και τα στατιστικά στοιχεία ποιοτικά. Και μια τελευταία ερώτηση θέσατε. Γιατί υπέβαλα αίτημα για αυτή την ε, θέση, για αυτό το αξίωμα. Όπως προανέφερα πολύ σύντομα, να πω επ' αυτού, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μοναδικό χαρακτήρα για το ότι δηλαδή ποιο ρόλο διαδραματίζουν τα στατιστικά στοιχεία και αποτελούν τη βάση πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται. Είτε είναι για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι για μέτρα και προτάσεις όπως 2-pack και 6-pack, τα διτά, διπλά μέτρα και ε, εξαπλά, εξαπλές διατάξεις. Αυτός είναι ένας λόγος. Αλλά στατιστικά και η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων και η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι πολύ χαμηλή δυστυχώς στην Ευρώπη η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά τα στοιχεία. Και αυτό εφαρμόζεται εφαρμόζεται, ισχύει για χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και όχι για κάποιες λίγες χώρες. Αν συναθλιστούν αυτά τα δύο στοιχεία, είναι πολύ σημαντικά λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία για την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπάρχει πολύ χαμηλή αξιοπιστία από πλευρά των πολιτών σε αυτά τα στοιχεία και χαμηλή εμπιστοσύνη. Δεν είναι λοιπόν υψηλή εμπιστοσύνη σε αυτά του πολίτε μα. Αυτό είναι ένα στοιχείο, στατιστικά στοιχεία βέβαια, αλλά πρέπει να δούμε γενικότερα σε ένα μεγαλύτερο εύρο τη σπουδαιότητα των στατιστικών στοιχείων. Θέλω λοιπόν να βελτιώσω τα πράγματα, να μπορέσουν να βελτιωθούν. Γι' αυτό υπέβαλα την αίτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος για την Άλντε. Yes. Ε, thank you, Chair. Εις παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό το ότι ήρθατε εδώ ενώπιόν μας. Καμιά φορά πιστεύει κανείς ότι είμαστε, θα έλεγε κανείς, ε, διανοούμενοι και στενόμυαλοι όσον αφορά την αυστηρή εφαρμογή κανόνων και κανονισμών. Όμως σε σχέση με τις ε, δραστηριότητες μιας κοινοβουλευτική ε, επιτροπής, ε, ποια θα ήταν η απάντησή σας στην κατηγορία ότι υπάρχει ιδιαίτερη αυστηρότητα και υπάρχει μονόπλευρη, μονοβαρής θα έλεγα επικέντρωση σε διάφορες δράσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, απαντά ο κύριος Χετεμέκη. Θα απαντούσα και θα έλεγα ότι και αυτά τα οποία έλεγα επ' αυτού είναι το εξή. Είναι τα εξής είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε σίγουρα. Δηλαδή ποιότητα και εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων. Δεν είναι το να είναι κανείς αυστηρός αυτό. Απλά αυστηρός. Είναι κάτι το οποίο είναι η απέτηση των πολιτών. Το διεκδικούν οι πολίτες και το απαιτούν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε καλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία για την λήψη πολιτικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι ελάχιστες απαιτήσεις για αυτά τα στοιχεία. Εσείς λαμβάνετε τις αποφάσεις βέβαια και πρέπει να έχουν υψηλή, υψηλό βαθμό ποιότητα σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία για να είναι σωστές, ορθές οι απαιτήσεις σας. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό θα έλεγα αυτό. Πρέπει να ισχύει. Thank you. Σας ευχαριστώ. Η Μαρίζα Ματίας από πλευρά της Ενωτικής Αριστερά. Το βριάδα. Ευχαριστώ. Κύριε Γεταμάκη, ευχαριστούμε. Ε, δεν μιλάμε με αφηρημένο τρόπο για τα στατιστικά στοιχεία και συμφωνώ μαζί σας πόσο σημαντική είναι η αποτίμηση διότι υπάρχουν πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά αυτές βασίζονται από τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από διάφορους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Eurostat. Ε, δεν πρόκειται όμως μόνο για σφάλματα στα στατιστικά στοιχεία. Το θέμα είναι η συγκρισιμότητα επίσης των στατιστικών στοιχείων και υπάρχει ένα συγκεκριμένο στατιστικός δείκτης ε, για τον, που είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος και θέλω ε, την άποψή σας. Νομίζω δικαιούμαστε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας. Γι' αυτό μιλώ για το για το διαρθρωτικό έλλειμμα και υπάρχουν ε, πολύ διαφορετικοί τρόποι μέτρησης του. Δεν υπάρχει ε, ε, μία μόνο μεθοδολογία για τον υπολογισμό του. Υπάρχουν ε, δύο διαφορετικοί τρόποι και στο δεύτερο λαμβάνεται υπόψη το καθάριστο εγχώριο εισόδημα. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι ιδιαίτερα υψηλή ανεργία 15% ή 30% σε μία χώρα και φαίνεται σαν μία τάση στην στατιστική αποτίμηση ενώ πρόκειται για βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ε, εάν ε, ε, υπάρχει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και δεύτερον, που επίσης είναι σημαντικό για την καθημερινή ζωή των πολιτών, υπάρχουν διάφορες εκδοχές ε, του, του δίκτυ. Δεν θέλω να σας κάνω μια εύκολη ερώτηση, θα ήθελα την άποψή για αυτό το δύσκολο ερώτημα. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μια ερώτηση η οποία δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΣΓΑΠ, αλλά επειδή και εγώ ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και βρίσκομαι εδώ ε, και είπα και στον πρόεδρο πριν από τη συνεδρίαση ότι έχω γράψει και σχετική εργασία επί του ζητήματος. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και να σας πω λοιπόν δύο λόγια από αυτού. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ε, ε, μέτρηση του διαρθρωτικού ελλείμματος και το θέμα είναι πώς η διαφορά μάλλον έγινε στο πόσο καθένας μετρά ε, το δυνητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε και κυκλικές μεθόδους διαρθρωτικής ισορροπίας. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, αλλά ε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Είναι κάτι όμως το οποίο ε, προτείνω να το εξετάσει η Επιτροπή σας ε, περαιτέρω. Συγγνώμη που είμαι τόσο σύντομη στην ερώτησή μου. Συγγνώμη. Έχετε όμως κάποια προτίμηση σε σχέση με τις μεθοδολογίες. Ε, η απάντηση ναι, έχω. Και αυτή είναι προσωπική άποψη βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με την ΕΣΓΑΠ. Προτιμώ περισσότερο την προσέγγιση που χρησιμοποιεί το Κογκρέσο, το, ε, η Υπηρεσία Προπολογισμού του Κογκρέσου. Χρησιμοποιεί μια διαρθρωτική μέθοδο και αυτό προϋποθέτει ότι ο τρόπος μέτρησης ε, του δημοσιονομικού ελλείμματος δεν εξαρτάται από τον κύκλο, είναι κάτι πολύ πιο σταθερό και ο κίνδυνος στη στατιστική μέθοδο είναι ότι μπορεί να έχουμε ε, μια προκυκλική αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ε, συζητηθεί πολύ περισσότερο και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ βέβαιος ότι και η εισηγήτρια για την αναθεώρηση της ε, ε, διακυβέρνησης θα ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η κυρία από τους ο κύριος Βανγκίκολ, συγγνώμη, με τους πρασίνους. Καλωσορίσατε και από πλευράς μας. Συμφωνώ, εμένα δεν μου αρέσει μόνο η φιλανδική πειθαρχία, αλλά και το φιλανδικό χιούμορ. Ε, το κράτος όμως που θεωρείται το πιο πειθαρχημένο και είναι πολύ πειθαρχημένο όταν πρόκειται για αριθμητικά στοιχεία, μπορείτε να δείτε ότι δεν ισχύει αν δείτε τι γίνεται στο αεροδρόμιο του Βερολίνου ή σε... Ε, εγκαταστάσεις ε, κατασκευής ε, πυρηνικών ε, σταθμών όπου δαπανούμε πολύ περισσότερα από όσα είχαμε προγραμματίσει και αυτό μάλλον δεν είναι και πολύ φιλανδικό. Τέλο πάντων αυτό ήταν απλή μια παρατήρηση. Έχω μια παρατήρηση, μια ερώτηση για τον οργανισμό τον οποίο θα αναλάβετε κανόνες για τον υπολογισμό ελλείμματος και χρέους και τα στατιστικά στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη επινοούν πάρα πολλούς τρόπους προκειμένου να αποκρύψουν το χρέος και το έλλειμμα. Ακόμα και ο κύριος Γιούγκερ έχει τη δική του εκδοχή τώρα. Αν ε, βάλει κάποιος χρήματα στο ε, επενδυτικό του κεφάλαιο δεν θεωρείται ότι είναι χρέος και έλλειμμα αυτό. Αν αναλάβει λοιπόν κάποιους κάποιους κινδύνους ε, υπό τη μορφή σιωδών λογιστικών αυτά δεν δεν συνυπολογίζονται. Επομένως θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, η Επιτροπή σας θα μπορέσει να συνεισφέρει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, σε αυτές τις ε, κινήσεις του χρέους και του ελλείμματος υπό μορφή σκιωδών λογιστικών και πώς μπορούμε να προβάλλουμε περισσότερο συγκεκριμένες ευθύνες, οι οποίες ε, είναι αυτές οι οποίες καλείται στη συνέχεια να καταβάλει ο λαός, αλλά τελικά φαίνεται ότι μέχρι τώρα ε, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να, λάβει τις ευθύνες. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Yeah, thank you, Mr. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολ. πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, όμως εκφεύγει ελαφρώς του πεδίου αρμοδιοτήτων της ΕΣΚΑΠ, παρότι ένας από τους στόχους είναι να ε, υποβάλουμε εκθέσεις για, τα, για την εκπόνηση στατιστικών στοιχείων και την τήρηση του κώδικα. Οπότε, απαντώντας, πρώτα να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και δεύτερον, οι κανόνες που έχουμε είναι φυσικό να επηρεάζουν αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις. Κάνετε και λαμβάνετε αυτό που μετράτε ε, τρόπον την Μιλήσατε για στοιχεία του παθητικού ε, που δεν εγγράφονται ε, και δεν καταγράφονται στο χρέος και, ότι, και λέτε ότι αυξάνεται ο αριθμός τους. Τα στοιχεία του ενεργητικού των ε, κυβερνήσεων που μειώνουν το καθαρό χρέος ε, βρίσκονται από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα. Υπάρχουν και οι δύο πλευρές, και τα στοιχεία του υποθετικού και του ενεργητικού. Ε, μόνο έτσι μπορεί κάποιος να έχει ρεαλιστική εικόνα για το ισοζύγιο. ή μάλλον για τον ισολογισμό, για τον προπολογισμό του κράτους. Ε, πρόσφατα ε, ε, δημοσιεύσαμε μία μελέτη όπου πραγματευόμασταν ακριβώς το θέμα του καθαρού χρέους και εκεί μιλήσαμε για το κρόστετ και για τα στοιχεία του παθητικού, τα άρετα στοιχεία του παθητικού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία απαντήσεων εκεί. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν από το EFTD. Η Μπάρμπαρα Κάπελ από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην ετήσια έκθεση η ΕΣΓΑΠ σε σχέση με την ε, διακυβέρνηση λέει σε σχέση με την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια των εθνικών στατιστικών στοιχείων. Το είπατε αυτό ζήτημα στην αρχική σας παρέμβαση. Ερώτησή μου, ποια μέτρα θα λάβετε εσείς ως μελλοντικός πρόεδρος της ΕΣΓΑΠ, ώστε <clears throat> στον δεοντολογικό κώδικα πρακτικών στις παραμέτρους όσον αφορά την ανεξαρτησία και διαφάνεια στο εθνικό επίπεδο δηλαδή σε σχέση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να εφαρμόζονται καλύτερα οι διατάξεις. Και γενικά, ποια κίνητρα θα προσφέρει η ΕΣΚΑΠ στις Εθνικές Στατιστικές Αρχές ώστε πλεονάζον δυναμικό να μπορέσει να ε, αντιμετωπιστεί και να εξυγχρονιστεί το στατιστικό σύστημα των κρατών μελών. Και επιτρέψτε μου μια περαιτέρω ερώτηση για τον έλεγχο όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για την διαχείριση ποιότητας ανήκει και η εξέταση των στοιχείων αυτών κατά πόσον είναι αληθή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο κώδικας πρακτικών λοιπόν προτείνει κάποιες δυνατότητες, προσφέρει κάποιες δυνατότητες για να μπορεί να ελέγχεται ο βαθμός αξιοπιστίας και αληθότητας, αλήθειας αυτών των στατιστικών στοιχείων. Και τι προτίθεστε να κάνετε για να βελτιωθεί αυτό. Ευχαριστώ. you, Σε ευχαριστώ πολύ. Το όπλο, αν μπορώ να πω, της ΕΣΓΑΠ είναι τα πιθανά προβλήματα να δημοσιοποιηθούν, να γνωστοποιηθούν και να αναφέρουμε τα προβλήματα αυτά σε εσά, στη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚΟΝ, στο Ευρωπαϊκό δηλαδή Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο ταυτόχρονα. Και έτσι οι δυνατότητες που υπάρχουν για να ανοιχνεύσουμε προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε στα, στις εθνικές στατιστικές αρχές δεν έχει την ικανότητα αυτή ε, η ΕΣΚΑ. Πρέπει να βασιστεί στην ε, Eurostat για να δράσει. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει είναι να αναφέρει σε εσά και στο Συμβούλιο τα όσα έχει συμπεράνει και τα έχει διακριβώσει η Eurostat για τις ε, δυνατότητες για τον κώδικα πρακτικών. Αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει κανείς και να δημοσιοποιηθεί η κατάσταση. Και όπως είπα πιο πριν, εργαζόμαστε με βάση την ήπια νομοθεσία. Δεν εργαζόμαστε με βάση νομοθετικά δεσμευτικούς κώδικες πρακτικών. Και γι' αυτό είναι ακόμα περισσότερο σπουδαίο και σημαντικό όταν να χρησιμοποιείται η δημοσιότητα, ο δημόσιος χαρακτήρας, ο ανοιχτός χαρακτήρας, να δημοσιοποιούνται τα πάντα με εκθέσεις, ε, γνωμοδοτήσεις, ε, διακριβώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολιτικά υπεύθυνοι να μπορούν να δράσουν ώστε να λογοδοτούν ε, όσοι είναι υπεύθυνοι για τα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Η ΕΣΚΑΠ δεν είναι αστυνομικό όργανο και δεν έχει έτσι την ικανό, τις ικανότητες και δεύτερον δεν έχει και την, το κύρος ή την ε, εξουσία να κάνει κάτι. Μόνο μπορεί να αναφέρει τα προβλήματα που υφίστανται σε εσά, το Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μέκη Ευχαριστούμε τους συναδέφους για τις ερωτήσεις. Και τώρα θα έχουμε μια και κλεισμένων των θυρών σύντομη συζήτηση για τα αποτελέσματα της ακρόασης ε, σε σχέση με τα όσα έχουμε σχεδιάσει για αύριο. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Μέκη για την παρουσία του ανάμεσά μας σήμερα και τις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις μας. Uh, Καλό τώρα μόνο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να παραμείνουν στην αίθουσα. Οι άλλοι να αποχωρήσουν παρακαλώ. Όλοι οι άλλοι που δεν έχουν ε, αρμοδιότητα και εργασία μπορούν να αποχωρήσουν παρακαλώ.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 Okay, we can start. Λοιπόν, να, να αρχίσουμε. Προτείνω να γίνει μια πολύ σύντομη ανταλλαγή απόψεων, να δώσω το λόγο στους συντονιστές ή τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για να σχολιάσουν